εδρίασή μας και έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Καταρχάς ανακοινώνω τη συνέχιση της διακοπής σας συνόδου που είχε διακοπή στις 17 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνόδου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Δεν νομίζω να υπάρχουν σχόλια. Άρα θεωρούνται τα πρακτικά ως ε, εγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας δώσω, να κάνω τις ανακοινώσεις, σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η γραπτή δήλωση 89 κάθετο 2010 έχει συλλέξει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών και γι' αυτό έγινε κείμενο υιοθετημένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η δήλωση εντάσσεται στη μονομερή επαναφορά των απαιτήσεων ε, θεωρήσεων από τον Καναδά για τους Τσέχους.